Meine Damen und Herren, darf die Sitzung zum Tag. Κυρίες και κύριοι, άρχεται η συζήτηση για το σημείο 9 της ημέρησιας διάταξης, συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερβαϊντάν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, το έχει, ε, έχει συμφωνήσει στην αντίστοιχη διαδικασία του, ε, η συγκήτρια κυρία Γκέτεν Μάκη. Εκπνέει σε λίγες ώρες η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών, στις 6 ώρα ακριβώς. Και ε, αντίστοιχες συμφωνίες έχουμε με την ε, Γεωργία, Μολδαβία, Αρμενία και Ουκρανία. Αυτή η συμφωνία λοιπόν θα δώσει τη δυνατότητα στο Αζερβαϊτζάν να υπογράψει ένα μνημόνιο συνεννόησης για διάφορα κοινοτικά προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να συμμετάσχει. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι πρόκειται για ένα τεχνικό αμυγός έγγραφο που θα επιτρέψει σε μια σειρά θεμάτων τη συνεργασία και το διάλογο με τρόπο πιο εντατικό και ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαπροσωπικές επαφές. People to people. Αυτό θα πρέπει να φέρουμε στο προσκήνιο και λιγότερο άλλα ζητήματα Θα παρακαλέσω την κυρία Γιατεμάκη να μας ενημερώσει για την κατάσταση των πραγμάτων και να μας διαφωτίσει, την οποία δεν βλέπω κιόλα. Είναι εδώ η κυρία Γιατεμάκη. Α, εκεί πίσω μάλιστα. Γιατεμάκη. Πώς σας λένε ακριβώς. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο όνομα με τόσα umlaut και τόσες διφθόγκους. Πολύ ωραία το, το προφέρετε. Μα εδώ προσπαθεί να με παραπλανήσει ο πρόεδρος. Ο συμπρόεδρος, έχετε το λόγο. When we spoke in the... Όταν ε, μιλήσαμε για το, για το προηγούμενο θέμα, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, είπε κάποιος ότι είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Θέλω να σας πω ότι το Αζερβαϊτζάν είναι επίσης μια πολύ όμορφη χώρα. Το Μπακού είναι πολύ ωραία πόλη και ο κόσμος είναι ε, πολύ ζεστός όπως είμαστε και εμείς. Ορισμένες φορές μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα Αλλά σίγουρα ε, δεν είναι το Αζερβαϊτζάν πρωτοτυπία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να έχει θέματα προς επίλυση με διάφορες χώρες. Το σωστό είναι να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονές μας και αυτή είναι η προσπάθειά μας. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι τεχνικό το ζήτημα, όμως είναι και σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Διότι το Αζερβαϊτζάν είναι σημαντικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έχουμε μια συνολική και βιώσιμη συνεργασία ε, περιλαμβανωμένη της ενέργειας, των αντιτρομοκρατικών δράσεων, των επιχειρήσεων, των επενδύσεων, του πολιτισμού, της παιδείας, της εκπαίδευσης μεταξύ άλλων και της έρευνας βέβαια. Στόχος λοιπόν αυτού του πρωτοκόλου είναι να καθορίσει τους οικονομικούς και τεχνικούς κανόνες που θα επιτρέψουν στο Αζερβαϊτζάν να συμμετάσχει σε ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το, βαθμιακό, το ε, σταδιακό, με άνοιγμα των προγραμμάτων προς τις χώρες αυτές παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 ήδη και το 2007 το Συμβούλιο υιοθέτησε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι βασική συνιστόσα της πολιτικής ε, γειτονίας και στόχος είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα, η συνεργασία ε, στην βάση της πυραμίδας της κοινωνίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί σε διάφορα πεδία. Ανταλλαγές φοιτητών, έρευνα, καινοτομία, ε, ανταγωνιστικότητα. Όπως είπε και ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ, Τέτοιου είδους προγράμματα ήδη έχουμε με την Αρμενία, τη Γεωργία, την Μολδαβία και την Ουκρανία. Προσωπικός είμαι υπέρ αυτού του πρωτοκόλλου διότι θεωρώ ότι ενισχύει τις επαφές μεταξύ πολιτών, Ευρωπαίων πολιτών και πολιτών του Αζερβαϊτζάν. Είναι κάτι που αφαιρά, αφορά άμεσα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους πολίτες του Αζερβαϊτζάν. Αμφότεροι θα υποφεληθούν. Το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία θα πρέπει να είναι οι βασικές αρχές που θα διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλες αυτές τις χώρες ε, συμπεριλαμβανομένου του Αζερβαϊτζάν. Αυτά είναι αυτά που μου ζήτησε ο Πρόεδρος να σας πω ε, και συμφωνώ. Ευχαριστώ. <laughs> Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε τη συζήτηση για το Συμφωνία Πλαίσιο για το Πρωτόκολλο μεταξύ της Ένωσης και του Αζερβαϊτζάν. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ε, ποια πολιτική κατάσταση γνωρίζει η χώρα, η οποία είναι εξαιρετικά ανησυχή, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά ε, διότι το έχει ε, δηλώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένο. Στα τελευταία χρόνια η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει υποβαθμιστεί ιδιαιτέρως, αυτό είναι γεγονός. Του τελευταίου μήνε έχει κλιμακωθεί η κυβερνητική καταστολή, οι ε, συλλήψεις, οι συλλήψει και φυλακίσεις υπερμαχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν από λίγους μήνες η Λέιλα Γιούνους ήταν στη τελική υποψήφια για το βραβείο Ζαχάροφ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι και η πιο γνωστή περίπτωση, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Είναι στη φυλακή από τον περασμένο Ιούλιο, για πολιτικούς λόγους έχει διωχθεί, έχει υποστεί ε, βία μέσα στο κελί και η υγεία της έχει υπονομευθεί και επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες. Είναι ακόμα μία υπόθεση, ακόμα μία περίπτωση μεταξύ ε, πολλών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή τη δυναμική, να δίνουμε βραβείο σε ορισμένους για τον αγώνα τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μετά να ξεχνάμε όλους τους υπόλοιπους ή και αυτούς τους ίδιους επειδή υποτίθεται εξυπηρετούμε την ε, πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τις αξίες και τα συμφέροντα αλλά και τις καλές σχέσεις με, όλους αυτούς τους, με όλες αυτές τις χώρες. Επομένως, στο πρωτόκολλο δεν γίνεται αναφορά και πρέπει να το θυμίσουμε αυτό, ότι πριν από λίγους μήνες, το Σεπτέμβριο, υιοθετήσαμε ψήφισμα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν υπάρχει αυτό στο κείμενο, αλλά είναι ξεκάθαρο το τι λέει το ψήφισμά μας για τις σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν. Σημείο 11. Η έγκριση της υπογραφής συμφωνίας σύνδεσης με το Αζερβαϊτζάν θα εξαρτάται από το κατά πόσο ε, με ικανοποιητικό τρόπο ικανοποιούνται τα αιτήματα των υπέροχων ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό το ψήφισμα υπογράψαμε πριν από λίγου μήνε και όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά έχει χειροτερεύσει κιόλα από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα. Επομένω, αν θέλουμε να έχουμε συνοχή με το κριτήριο που έχει υιοθετήσει ε, σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ολομέλειά του, στο σχετικό ψήφισμα, θα πρέπει να είμαστε κατά της έγκρισης αυτού του πρωτοκόλου. Και ως εκ τούτου ε, θα υποβάλλουμε τροπολογία σχετική. Και όσο δεν βελτιώνεται το κείμενο ως προς τις αναφορές για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα θα είμαστε εναντίον και θα πρέπει να ε, θυμίσουμε την δραματική περίπτωση της Λέιν για να σώσουμε και τη ζωή της, διότι η υγεία της κινδυνεύει. Όλα αυτά ε, σχετίζονται με την καθημερινότητα, με τους καθημερινούς ανθρώπους που ζουν σε αυτή τη χώρα. Και θα πρέπει ε, να το λάβουμε υπόψη και την επόμενη φορά που θα, συζητήσουμε, θα συζητήσουμε για αυτό το πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, μετά τη συνεδρίαση θα σας παρακαλούσα να ενημερωθείτε για τη τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων και τις πρόσφατες εξελίξεις. Mrs. Η κυρία Σεμπάλιους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτά που είπε η κυρία Γιατεμάκη. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε ό,τι κάνουμε για την πολιτική αυτή. Ακούσαμε όμως και από τον Ισπανό συνάδελφο ποια είναι η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Είναι πολύ άσχημη και έχει επιδεινωθεί τους τελευταίους μήνες είναι κάτι που έχουμε παρακολουθήσει από κοντά. Ξέρουμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε τι υπάρχει και στην έκθεση. έκθεση η οποία δεν αντικατοπτρίζει όμως απόλυτα τη σημερινή κατάσταση. Τι μπορούμε να πούμε. Να αποφανθούμε όσον αφορά αυτή την έκθεση. Δίνουμε όμως ένα κακό μήνυμα. Η κατάσταση επιτόπου είναι πολύ άσχημη. και δεν συμφωνεί με το περισσότερα για περισσότερα. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να αναβάλουμε την εξέταση αυτού του θέματος, ίσως και μερικούς μήνες. Ίσως αργότερα να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει επί τόπου όσον αφορά κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Πακού και γενικότερα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Το Αζερβαϊτζάν παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παίξει και ακόμα πιο σημαντικό. Μια που θέλουμε και εμείς τον διάδρομο φυσικού αερίου. Πρέπει να προσέξουμε τι υπογράφουμε και τι θέλουμε. Το Αζερμπαϊτζάν έχει μια δικτατορία με πολιτικούς κρατούμενους. Σλάζοβα για παράδειγμα που έχει συλληφθεί και κατηγορείται ότι έχει επηρεάσει άλλον ε, ρεπόρτερ εκεί. Το έγκλημά της με την γυναίκα είναι ότι ακριβώς έχει επηρεάσει το κλίμα στη χώρα. Επηρέασε να φτάσει και η σχετική έκθεση στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εμείς πρέπει να καταδικάσουμε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Το εμπόριο με το Αζερβαϊτζάν θα πρέπει να εξαρτηθεί από την απελευθέρωση κρατουμένων όπως είναι αυτός στον οποίο αναφέρθηκα πριν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπε ο σκιώδης εισηγητής μας, λέει η κυρία Πύρη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση που πηγαίνει σε ΜΚΟ ε, που ελέγχονται από την κυβέρνηση. Δεν είναι ο λαός προς το λαό. Έχουμε ανοίξει ε, αυτά τα κονδύλια ε, για ελεγχόμενες από την κυβέρνηση οργανώσεις, ενώ οι πραγματικοί αγωνιστές φυλακίζονται ένας μετά τον άλλο. Η Λευκορωσία δεν έχει συμφωνία ε, μαζί μας για αυτό το λόγο και δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι πολυκριτικοί κρατούμενοι στο Αζερβαϊτζάν από ότι είναι στη Λευκορωσία. Αυτό μας κάνει να σκεφτόμαστε την κατάσταση. Κοιτάξτε, δεν έχουμε άλλα θέματα. Η συμφωνία πλαίσιο είναι μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερβαϊτζάν. Θέλει κανείς άλλο το λόγο γι' αυτό. Α, η κυρία Γιατεμάκη προφανώς η συγγήτρια για να κλείσει. Madame rapporteur. Some questions. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι εδώ δεν πρόκειται για συμφωνία σύνδεσης με το Αζερβαϊτζάν. Μπορεί αυτό να συμβεί αργότερα, δεν ξέρω. Εδώ πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα που βοηθάει τον κάθε πολίτη του Αζερβαϊτζάν και η δικιά μας η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συμφωνία αυτή όμως ακριβώς προσπαθεί να βοηθήσει τον κοινό κάτοικο του Αζερβαϊτζάν με ανταλλαγέ νέων, ώστε οι νέοι να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ή να σπουδάσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να μάθουν ακριβώς τι σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα και τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρόκειται για συμφωνία σύνδεσης. Και το γνωρίζω ότι υπάρχουν προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αζερβαϊτζάν. Όλοι μας το ξέρουμε. Αλλά ακόμα και αν υπάρχουν, πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον καθημερινό άνθρωπο, τον κοινό άνθρωπο στο Αζερβαϊτζάν να ενημερωθεί καλύτερα, μελετώντας ή επισκεπτόμενος ευρωπαϊκές χώρες και ανάποδα. Αν και εφόσον υπάρξει συμφωνία σύνδεσης, αυτό θα είναι άλλο θέμα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα τότε. Και δεν μπορώ, δεν ξέρω πότε θα προκύψει και αν θα προκύψει. Τώρα όμως έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα μπροστά μας προκειμένου να βοηθήσουμε τους απλούς κατοίκους του Αζερβαϊζάν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία εισηγήτρια, κυρία Γιάτεμάκη. Και όντως είναι μια σημαντική συμφωνία πλαίσιο η οποία θα βοηθήσει το Αζερβαϊτζάν να ενισχύσει τις επαφές ε, μεταξύ των ανθρώπων από το Αζερβαϊτζάν και την Ευρώπη. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι αύριο, 1η Απριλίου, στις 3 το μεσημέρι. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, Ευχαριστώ την εισηγήτρια και ολοκληρώνουμε έτσι το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να ενημερωνόμαστε για να μην βλάπτουμε ε, με καλές προθέσεις τελικά να, ε, να έχουμε το αντίστροφο αποτέλεσμα. Καμιά φορά οι καλές προθέσεις είναι ο εχθρός του καλού. Έτσι, οι καλές προθέσεις μπορεί να βλάπτουν καμιά φορά κιόλα. Πάμε λοιπόν στο σημείο 10. Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν. Κυρία Λέζεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήδη με email έχουν ε, προηγηθεί ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των σκιωδών εισηγητών για την έκθεσή μου που έχω καταθέσει. Πρέπει να σας πω ότι το βρίσκω ασυνήθιστο κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα να θυμίσω την κανονική διαδικασία και να ακολουθήσουμε ε, τους δημοκρατικούς κανόνες και να συζητήσουμε κανονικά την έκθεσή μου. Οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων συζητούν εδώ και με διαφάνεια και εδώ θα πρέπει να γίνεται η πραγματική ανταλλαγή απόψεων και όχι σε διάφορα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Μα γι' αυτό σας έδωσα το λόγο, για να γίνει αυτός ο διάλογος. Τι συζητάτε τώρα, λέει ο πρόεδρος που διακόπτει την ομιλήτρια. Ναι, θέλω να πω όμως τι συνέβη. Ορισμένοι σκιώδοι συζητητές εκ των προτέρων προσπάθησαν να στείλουν email για να κάνουν τη συζήτηση γραπτός. Μα δικαίωμά τους είναι. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω και τη χαρά μου που συμφωνείτε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε εδώ. Και λίγη αυτή η ιστορία. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά δεν κατάλαβα την αιτίασή σας. Οι συνάδελφοι έχουν πάντα το δικαίωμα πριν, μετά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να στέλνουν και mail και ό,τι άλλο θέλουν. Εντάξει, τώρα θα τσακωθούμε γι' αυτό. Ε, λέτε να μην το συζητήσουμε. Αυτό δεν το συζητάω αυτό το διαδικαστικό. Χαίρομαι λοιπόν που όπως αρμόζει το συζητούμε εδώ δεν είναι ούτε αιτιάσεις, ούτε κρίσεις, ούτε αξιολογήσεις. Λοιπόν, η έκθεσή μου. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δυνατόν, δεν ξέρω, είναι σπάνιο σε τέτοιες εκθέσεις, να αναφέρουμε συνολικά όλα τα στοιχεία που αφορούν μια χώρα. έχουμε τεχνικές προδιαγραφές της γραμματείας και αναγκάστηκα να περικόψω κάπως την πρώτη μου εκδοχή και έχω κρατήσει μόνο τις, τα μεγάλα κέντρα βάρους. Και θα ήθελα να σας αναγγείλω ήδη ότι θα κάνω τροπολογίες για όσα δεν μπόρεσα να χωρέσουν στην έκθεση για να τις συμπληρώσω. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τη γραμματεία για την συνεργασία μας έχουμε διαφωνία. Ε, αυτό το έχουμε ακούσει επανειλημμένως ε, με ε, τις στρατιωτικές επεμβάσεις. Καταρχήν είμαστε αντίθετοι. Εμείς ως η αριστερά, η Λίνκε της Γερμανίας αλλά και το ειρηνευτικό κίνημα από την αρχή θεωρούσαμε ότι στα Αφγανιστάν ήταν λάθος η στρατιωτική επέμβαση. Ιδιαίτερα τα δικαιώματα των γυναικών ε, πλήττονται ε, πολύ και δεν μπορούν να εφαρμοστούν ούτε αυτά ούτε μια δυτικόστροφη κοινωνία. Δεν ήταν αυτό όμως που με οδήγησε να κάνω την έκθεση, αλλά βασίστηκα σε εκθέσεις κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εμπειρογνωμόνων, διάφορα έγγραφα, τεκμηρίωση από φορείς, ε, από εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης και αυτά με οδήγησαν τα συμπεράσματα που έχω καταθέσει. Ότι θα πρέπει να δοθούν νέα βήματα να αναλυφθούν για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος της βίας. και μόνο το έτος 2014 είχαμε από άμαχο πληθυσμό θύματα 10.548 παρακαλώ. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τις προσπάθειες και τις επιτυχίες ε, που έκανε η χώρα για την ανοικοδόμησή της. Δεν θέλω να το υποτιμήσω καθόλου. Αλλά και από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει εμείς να αξιολογήσουμε την πραγματική κατάσταση, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να προτείνουμε ε, κάποια σημεία για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. εγώ βασίζομαι σε μια προσεκτική διαβούλευση όσο γίνεται ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων, είπαμε ΜΚΟ και άλλων φορέων έχουν εμπλακεί. Θα παρακαλούσα κάπως τους συναδέλφους να μην κάνουν τόση φασαρία για να μπορέσω πιο εύκολα και πιο γρήγορα να σας παρουσιάσω την έκθεση. Η διαβούλευση δεν τελείωσε με την υποβολή της έκθεσης, ακόμα και όταν τελείωσα το γράψιμο και την κατάρτισή της, ε, ήρθα σε επαφή με εκπροσώπους της Διεθνούς Διαφάνειας, για την διαφθορά ή για το Human Rights Watch για τα βασανιστήρια και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με μια τιμωρησία που διαιωνίζεται και που γίνεται ε, ανεκτή. Θα κάνω και τροπολογίες σχετικά. Σύντομα θέλω να πω κάτι ε, απαντώντας στην επιστολή του Αφγανού πρέσβη ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι είναι η έκθεσή μου κάτι το οποίο τον ανησυχεί και τώρα που αναλαμβάνει η νέα κυβέρνηση δεν είναι σκόπιμο και τον λυπεί. Αλλά σας είπα και μετά από συνεννοήσεις με διαφόρους και με το Human Rights Watch ε, μου είπαν ότι είναι ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε, να δράξουμε αυτή την ευκαιρία του σχηματισμού της νέας κυβέρνησης για να μπουν νέα ορόσημα και νέα θεμέλια. Νομίζω ότι είναι πρόσφορο το έδαφος και ο καιρός είναι ευκαιρία για να βάλουμε κάποια benchmarks να τα εφαρμόσουν ιδιαίτερα για τη διαφθορά, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γυναικείων δικαιωμάτων και να μην υπάρχει αυτή η διαρκής ατιμορρησία. Στην έκθεσή μου συνδέω τη φτώχεια με τη ριζοσπαστικοποίηση και χρειάζεται οπωσδήποτε να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Η μαζική ανεργία επίσης είναι ζήτημα 50% περίπου του συνόλου της ανεργίας. Κάθε χρόνο 400.000 νέοι μπαίνουν στην ε, ανεργία. Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση. Η συνέχιση ε, των ε, μαθημάτων στο σχολείο, ιδιαίτερα τα κορίτσια, και δεν το αμφισβητώ καθόλου αυτό, έχουν βελτιωθεί και τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών, αλλά αν δείτε ποια τεράστια πρόκληση έχουμε ακόμα μπροστά μας, θα καταλάβετε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Και θα πρέπει να κρίνουμε και τα όσα έχουν γίνει με βάση τα μέσα και τους πόρους και τα χρήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, πρόβλημα με την καλλιέργεια παπαρούνας ε, και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι αναπτυξιακή βοήθεια και ε, ανθρωπιστική αηφόρος για μια βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας και μια ανεξαρτησία τελικά ως μακροπρόθεσμο στόχο. Και συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. Άλλα σημαντικά στοιχεία και πάλι το θέμα της συνεργασίας στρατού και πολιτικών δυνάμεων, μη στρατιωτικών, και αυτό δεν το έχω βγάλει από το μυαλό μου. Τελειώνω, πρόεδρε, τελειώνω. Ναι, να τελειώνεται όμως. Έχω συναντηθεί με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων και με τα τεχνικά συνεργεία αντιμετώπιση καταστροφών, τα διάφορα σωστικά συνεργεία. Τα έχω βάλει όλα αυτά στην έκθεση. Τέλος, μία πρόταση. Το Αφγανιστάν είναι μια πλούσια χώρα με ένα εξαιρετικά φτωχό πληθυσμό. Άρα θα πρέπει να αναρωτηθούμε πώς είναι δυνατόν ο πλούτος αυτός να μην φτάνει στους ανθρώπους για μας είναι τεράστια πρόκληση. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα αλλάξει όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και πάλι να διαπιστώσω ότι δεν ήταν αυθαιρεσία της γραμματείας σε όλες τις εκθέσεις του Κοινοβουλίου έχουμε κάποιους κανόνες ως προς το μήκος τους και την έκτασή τους. Δεν ε, είναι κάτι που έχει να κάνει με τη δική σας ειδική περίπτωση. Είναι γενικός κανόνας και θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να καταλάβουμε ότι και στην Ολομέλεια αυτές θα πρέπει να μπορούν να ε, ψηφίζονται. Δεν είναι έκθεση ιδεών τι θεωρούμε σωστό ή λάθος, χωρίς ε, περιορισμούς. Το ψήφισμα είναι περιορισμένο, καταλαβαίνετε. Σε μια, ένα μηχανισμό και μια μηχανή όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο. Τώρα, η συζήτηση. Ο κύριος Ντανζόν. Παρακαλώ να είμαστε όλοι σύντομοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος εξ του ΕΛΚ. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με αυτή την έκθεση. Αναφέρεται ρητό στο άρθρο 1 ένας ε, ιδεολογικός διάβλος, ότι δηλαδή όλα τα δεινά του Αφγανιστάν προέρχονται από τη διεθνή στρατιωτική παρέμβαση του ε, Σεπτεμβρίου του 2001. Αυτό είναι μία απλούστευση που δεν μας επιτρέπει να έχουμε αντικειμενική θεώρηση της ε, κατάστασης και άρα καθίσταται προβληματική όλη η ανάπτυξη των ιδεών της έκθεσης. Μπορεί κανείς να ζητήσει τα δεινά και τα πλεονεκτήματα της ε, διεθνούς στρατιωτικής παρέμβασης στο Αφγανιστάν, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες. Είναι, έτσι έχουμε ε, feedback αν θέλετε. Είναι κάτι που γίνεται ε, από ε, τις στρατιωτικές δυνάμεις ούτως ή άλλως και είναι απολύτως θεμητό. Όμως εξ αρχής να λέμε ότι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έσφαλαν ε, μόνο μιας με την στρατιωτική διεθνή παρέμβαση στο Αφγανιστάν συνολικά είναι κάτι που δεν μπορεί να είναι δεκτό έχουμε οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία. Αυτά είναι νούμερα που δίδονται έτσι εν θερμό, ε, δηλαδή ε, παίρνονται μεμονωμένα και δεν μπαίνουν στη σωστή προοπτική. Υπάρχει δηλαδή ασυνέπεια. Από τη μία έχουμε δύο παραγράφους που εξηγούν ότι τα διεθνή κονδύλια δεν πρέπει να πάνε στο σκέλος της ασφάλειας αλλά στο σκέλος της ανάπτυξης και από την άλλη λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεσμεύεται περισσότερο για να χρηματοδοτήσει το στρατιωτικό σκέλος και να βοηθήσει στην ασφάλεια των Αφγανών ε, πολιτών, του Αφγανικού λαού. Υπάρχει λοιπόν ασυνέπεια μεταξύ αυτών των δύο διατυπώσεων. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικές ομάδες θέλουν να ε, ε, τροποποιήσουν ουσιαστικά ε, την έκθεση αυτή. Δεν είμαι, σίγουρη ότι θα τα, δεν σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε, ειδικά με τις στενές προθεσμίες που έχουν τεθεί. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η κατάσταση είναι πολύ ευμετάβολη, μεταβλητή στο Αφγανιστάν. Επομένως είναι μεγάλη πιθανότητα αυτό που, θα γράψουμε και θα εγκρίνουμε σήμερα π.χ. να είναι τελείως εκτός πραγματικότητας σε ένα μήνα είτε προς τη μία ε, κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Άρα το κατά πόσο αξίζει και είναι σκόπιμο να έχουμε ψηφοφορία ψήφιση τέτοιου είδους ε, ε, έκθεσης τους επόμενους δύο μήνες είναι κάτι που είναι απολύτως τυχαίο. Θα πρέπει, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου να το μεταθέσουμε χρονικά για αργότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι και εμείς διαφωνούμε με την έκθεση αυτή. Γιατί κατά τη γνώμη μας ξεκινάει από μια λάθος βάση, ότι δηλαδή η δυτική στρατιωτική παρέμβαση στο Αφγανιστάν ήταν ένας παράγοντας ριζοσπαστικοποίησης όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και οδήγησε στην αστάθεια στο Αφγανιστάν. Δεν είναι η άποψή μας. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να συζητήσουμε επί μακρό όσον αφορά τα υπέρ και τα κατά των διαφόρων δυτικών παρεμβάσεων που κατά τη διάρκεια ολόκληρη τη ιστορία έγιναν αισθητέ στο Αφγανιστάν και όχι μόνο. Να συζητήσουμε πότε ήταν αρνητικέ οι παρεμβάσεις αυτές και πότε θετικέ. Πιστεύουμε πάντως ότι η έκθεση αυτή βασίζεται σε αυτό το λάθος ήδη από την εκκίνηση και καταλήγει σε μια ιδεολογική ε, περιγραφή της πραγματικότητας. Η περιγραφή του Αφγανιστάν στην έκθεση αυτή είναι κάτι που δεν μας ικανοποιεί καθόλου και ο πρέσβης του Αφγανιστάν παρενέβη μάλιστα για να επιστήσει την προσοχή του συγητή στο γεγονός ότι η έκθεση αυτή απομακρύνεται πολύ από τα πραγματικά σημερινά συμφέροντα του Αφγανιστάν και ο ίδιος ο πρόεδρος του Αφγανιστάν πριν από μερικές μέρες στην Αμερικανική Γερουσία είπε ότι ήθελε οι δυτικές στρατιωτικές δυνάμεις να παραμείνουν περισσότερο στο Αφγανιστάν. Και μάλιστα εξέφρασε και την ικανοποίησή του για την ε, διαθεσιμότητα που έδειξε η Δύση. Γνωρίζουμε την κατάσταση. Πέρα από την εκτίμηση του καθενός για το κατά πόσο καλός ή κακός ε, είχαμε παρέμβαση στο Αφγανιστάν, το να πάρθει βιαστικά η απόφαση απόσυρση από το Αφγανιστάν είχε αρνητικέ συνέπειε στη χώρα γιατί δεν υπήρχε σταθερότητα, ούτε ειρήνη, ούτε προοπτική για λύση των προβλημάτων. Αντίθετα, αποτελεί ένα στοιχείο αστάθεια και χειροτερεύει η κατάσταση. Χειροτερεύουν ε, η φτώχεια και η μιζέρια στη χώρα. Μπορούμε να το συζητήσουμε ή όχι εδώ. Αυτό Μπορούμε να τον ερωτηθούμε, αλλά η ρευστότητα, η αστάθεια είναι πράγματα που δεν μπορούμε να τα πούμε οριστικά. Η κατάσταση αλλάζει από μέρα σε μέρα. Δεν μπορούμε δογματικά να το πούμε. Υπάρχει μια έκθεση του Κοινοβουλίου για το Αφγανιστάν και ένα κείμενο πάνω στο οποίο υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες αξεπέραστες για θέματα βασικά που αναφέρονται στην έκθεση η οποία αναλύει την κατάσταση στο Αφγανιστάν με τρόπο με τον οποίο δεν συμφωνούμε καθόλου. Τελειώνω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι η άποψη αυτή είναι άποψη πολύ ιδιαίτερη της Δύσης και πολύ αρνητική όσον αφορά την παρέμβαση της δύση στο Αφγανιστάν. Δεν είναι αποδεκτή, αλλά δεν σημαίνει βέβαια ότι το θέμα αυτό δεν πρέπει να συζητηθεί. Το είπε και προλαλή σα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί, αλλά βάση, με μια βάση διαφορετική, από ένα διαφορετικό σημείο κίνησης. Uh, thank you very much, Chairman. Well, I... Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει ο κύριος Βαν συμφωνώ πολύ με του δύο προηγούμενου ομιλητέ. Θα είμαι πολύ σύντομο. Έχω την εντύπωση ότι η έκθεση έτσι όπως έχει διατυπωθεί ε, ακολουθεί ιδεολογικό αντιαμερικανισμό, αντιστρατιωτικές τάσεις εξ αρχής. Και αυτό διαπνέει όλα τα επιχειρήματα που προβάλλονται. Μπορώ να σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα ανακριβιών που αναφέρονται σε γεγονότα που δεν έχουν συμβεί, που είναι λάθος. Για παράδειγμα, στην πρώτη παράγραφο λέγεται ότι μετά από 13 χρόνια δυτικής παρέμβασης έχουμε 10.548 παιδιά που έχουν για παράδειγμα τραυματιστεί. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, οι εξεγέσεις, ε, οι ε, μέσα στη χώρα ήταν αυτές που οδήγησαν το 72% των απολειών ε, ούτως ή άλλως. Στη δεύτερη παράγραφο καλούνται τα ΙΠΑ και το ΝΑΤΟ να αποσύρουν ε, το στρατιωτικό τους προσωπικό από τη χώρα. Η, η πραγματικότητα είναι άλλη. Έχει επιβραδύνει το ρυθμό απόσυρσης ε, στράτιωτων το κράτος των ΗΠΑ μετά από συγκεκριμένο αίτημα του Προέδρου Γκάνη. Στην παράγραφο 11 Αναφέρεται η έλλειψη ουσιαστικής πρόοδου σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στις γυναίκες και στα κορίτσια στο Αφγανιστάν. Όμως, το γεγονός παραμένει ο αριθμός των κοριτσιών που πηγαίνουν σχολείο στο Αφγανιστάν ταν έχει αυξηθεί από το 3% στο 36% σήμερα. Πάνω από 3 εκατομμύρια ε, κορίτσια Αφγανές πηγαίνουν στο σχολείο ενώ δεν πήγαιναν πριν. Στην ε, παράγραφο 14. Άλλη ανακρίβεια είναι η εξή. Λέγεται ότι όλα τα κονδύλια πρέπει να πηγαίνουν στην ανάπτυξη και όχι στην ασφάλεια. Να σας ρωτήσω λοιπόν το εξής. Η εκαθάριση ναρκοπαιδείων Πώς ταιριάζει η εξουδετέρωση των αρκών ε, με αυτό το επιχείρημα. Ε, μισό εκατομμύριο δολάρια έχουν δαπανηθεί ε, μέσα σε μια χρονιά από τη ΣΥΠΑ για την αποναρκοθέτηση. Και πολλοί έχουν δεχτεί απειλές και έχουν διακινδυνεύσει. Ακριβώς λόγω του κινδύνου των ναρκοπαιδείων. Αν δηλαδή δούμε το, το κείμενο παράγραφο προς παράγραφο, ε, βρίσκουμε συνεχώς τέτοιου είδους παραδείγματα. Είναι μη αποδεκτό, ε, δεν θα πρέπει να χάσουμε χρόνο προσπαθώντας να το τροποποιήσουμε, θα πρέπει να αποσυρθεί και να επανασυνταχθεί, ε, επαναδιατυπωθεί. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. President. Dear Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του κ. Σταδίτσιος που είναι από την άλλη πρέπει να πω ότι λυπούμαστε αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε την έκθεση αυτή. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο έτσι όπως έχει μεροληπτεί όσον αφορά τη σημερινή πολιτική κατάσταση στο Αφγανιστάν. και αγνοεί τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Είμαστε πεπισμένοι ότι η παράγραφη 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 16 και 17 θα έπρεπε να διαγραφούν πλήρως και η υπόλοιπη έκθεση απαιτεί επαναδιατύπωση. Ο σκέτος εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να ξαναγραφεί η έκθεση ώστε να παρουσιάσει μια αμερόληπτη άποψη για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά. Λαμβάνοντα υπόψη την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών που είναι σύντομα, θέλουμε να σας ζητήσουμε να υπάρξει νέο σχέδιο έκθεσης. Ο κύριος Αστρεβίτσιος που συμμετέχει στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας και με άλλους συναδέρφους από άλλες πολιτικές ομάδες προκειμένου να έχουμε μια καλά ισορροπημένη έκθεση που να αντικατοπτρίζει την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο στο Αφγανιστάν. Σας ευχαριστώ. Κυρία ε, ε, ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων θέλω να πω ότι πιστεύουμε πως είναι καλό που εμφανίζεται τώρα η έκθεση αυτή. Είναι σωστή στιγμή να συζητήσουμε και την κατάσταση στο Αφγανιστάν και για το μέλλον του. Και αυτό γιατί έχουμε την αποστολή που λύγει τώρα και έχουμε και τη σχέση με την αποστολή Μανάσκου και την ΙΣΑΦ. Δεν πρέπει να υπάρχει παράλυση. Εγώ συμφωνώ ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για να λυθεί η κατάσταση στο Αφγανιστάν. Συμφωνούμε με πολλά από τα σημεία της κυρίας Λέσινγκ. Συμφωνούμε με αυτά, με μερικά μερικώς, αλλά είναι η δυνατότητα, υπάρχει δυνατότητα για μας να υποβάλουμε προτάσεις τροπολογίας για να πούμε με τι συμφωνούμε και με τι συμφωνούμε. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή όλοι και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα για να προσφέρουμε και τις δικές μας απόψεις. Η κυρία Λέσινγκ αναφέρθηκε επίσης με την Transparency International και τις συναντήσεις με άλλες ομάδες και αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που γίνονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπογραμμίζω ότι και εμείς πρέπει να δουλέψουμε για το Αφγανιστάν. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην ειρήνη μακροπρόθεσμα, όχι μόνο πώς να σταματήσει βραχυπρόθεσμα η, η συγκρούση, αλλά να φροντίσουμε να μπορούν οι κάτοικοι εκεί να ζήσουν με ειρήνη και με δημοκρατία. Τώρα, για τις πολιτικές δυνάμεις, στρατιωτικές δυνάμεις κτλ. Όντως πρέπει να ανταμειχθούν. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα πλαίσια. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε και άλλοι να περάσουν από την αστυνομία σε εγκληματικές οργανώσεις. Οι παράγοντε αυτοί πρέπει να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους. Να μπορούμε και να συνεργαστούμε επίσης με κινήματα των πολιτών και ο πληθυσμό της χώρας να μπορεί να ζήσει βγάζοντας το ψωμί του τίμια από τη δουλειά του. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν το Αφγανιστάν να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, να υποβάλουμε τροπολογίες που να ικανοποιούν τις ομάδες μας. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να αναβάλουμε την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο, Πρόεδρος. Κυρία Λιωμαρή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν αμφιβάλλω ότι η κυρία Λέζινγκ διάβασε πολλά έγγραφα και είχε πολλές επαφές με διαφόρους. Προσωπικά έχω μεταβεί 14 φορές στο Αφγανιστάν, 14, όχι μόνο στην Καμπούλ και στο Κανταχάρ, Τζελαλαμπάτ, σε μεγάλες πόλεις αλλά και σε μικρά χωριά, πολύ μικρά χωριά και κοινότητες και έχω συζητήσει με αρκετούς και πάρα πολλές γυναίκες. Και μπορώ να πω το εξής. Σε αυτή την έκθεση δεν αναγνωρίζω τίποτα από όσα είδα εκεί. Τίποτα. Έχω δει ένα Αφγανιστάν το 2001, αρχές 2002 και είδα και τα όσα έχουν γίνει έκτοτε. Δεν είναι το θέμα καθόλου να πούμε ότι όλα είναι ρόδινα στο Αφγανιστάν, αλλά όταν μία έκθεση βασίζεται σε τόσα σφάλματα όσα η συγκεκριμένη, τότε δεν είναι σοβαρή απλούστατα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο τελικά χάνει ε, την ε, εικόνα του σε όσους το διαβάσουν και στο Αφγανιστάν. Πρέπει να σας πω ότι οι γυναίκες με τις οποίες συζήτησα δεν ε, ήταν κατά της διεθνούς στρατιωτικής επέμβασης που τις προστάτευσε και τους επέτρεψε να ξαναγυρίσουν σε σχολεία και σε γυμνάσια τα κορίτσια, διότι αυτό απαγορευόταν. Υπάρχουν κορίτσια που σκότωσαν οι Ταλιμπάν και γυναίκες γιατί προσπαθούσαν να διδάξουν σε κορίτσια για να μπορέσουν οι γυναίκες να απελευθερωθούν. Στο κοινοβούλιο εδώ λοιπόν έχουμε μια υποχρέωση και αυτή ποια είναι ηθική υποχρέωση, ηθικό χρέος να λέμε τα πράγματα και πράγματα σωστά, μετρημένα και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις και όχι απλά ε, ε, να έχουμε ε, ωραία λόγια και μεγαλόστομα που δεν οδηγούν πουθενά το Αφγανιστάν αξίζει να μιλάμε σοβαρά και να κάνουμε σοβαρές προτάσεις γι' αυτό. Um, Ο κύριος Καν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να μπω στη συζήτηση των υπέρ και των κατά το σαφές είναι ότι τα πράγματα στο Αφγανιστάν είναι πολύ χειρότερα τώρα από πλευράς βίας, διαφορά ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής από ό,τι στη δεκαετία του 70 και εν πάση πριν την ε, δική μας εμπλοκή και την ε, παρέμβαση τη διεθνή. Το παρελθόν μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το τι συμβαίνει στο Αφγανιστάν αλλά ε, πληρώνουμε το τίμημα όταν αγνοούμε την κατάσταση. Πρώτον, η σχέση Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι περίπλοκη. Τα σύνορα είναι μεγάλη έκταση, είναι δύσκολα και πρέπει να, πάει προς, πρέπει να προς μια καλύτερη κατεύθυνση η σχέση αυτή. Δεύτερον, η πληθυσμιακή ομάδα των Παστούν είναι πιο μεγάλη ε, στο Αφγανιστάν και πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία για να μην γίνει αυτό που έγινε και στο Ιράκ όπου οι Σουνίτες Άραβες δεν ενεπλάκησαν και αυτό ήταν ε, προβληματικό. Έχουμε δει στο παρελθόν πόσοι κίνδυνοι έχουν δημιουργηθεί από τη δράση των στρατιωτικών ομάδων και δεν θα πρέπει να επιδεινωθεί η κατάσταση από αυτή την έννοια. Ευχαριστώ. Επόμενος ο μιλητής. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τάνοκ. Οι Αμερικάνοι δεν παρενέβησαν ε, επειδή υπήρχε η δεκαετία του 70, παρενέβησαν γιατί η Αλκάιντα έκανε επίθεση στους δίδυμους πύργους και είχε την έδρα της στο Αφγανιστάν και γι' αυτό ε, υπήρξε η διεθνή στρατιωτική παρέμβαση. Συμφωνώ με τους συναδέλφους, η κυρία Λέζιν αρνείται πόσο έχουν βελτιωθεί τα δικαιώματα ε, των γυναικών στο Αφγανιστάν και αυτό μου προκαλεί μεγάλη έκπληξη από κάποιον που ανήκει στην Τιλίνκε. Η κυρία Λέσιν αγνοεί ότι οι Αφγανές γυναίκες λιθοβολούνταν μέχρι θανάτου ε, στο παρελθόν και πριν την παρέμβαση προτιμά αυτά τα μεσονικά, αυτή τη μεσονική κατάσταση, τουλάχιστον τέτοιου τους λιθοβολισμοί δεν γίνονται πια μετά την παρέμβαση του ΝΑΤΟ. Συμφωνώ με τον κύριο Βανόρντεν. Το μόνο που τη διαπνέει την κυρία Λαζίνη είναι οι αντιαμερικανικές απόψεις ε, και αυτό δεν μπορούμε εμείς να το δεχθούμε στο ECR. Ε, η Γκουε για άλλη μια φορά αγκαλιάζει την ειρηνική στάση, από την άλλη έχει κομμουνιστικά κόμματα που χειροκρότησαν την παρέμβαση της Σοβιετικής Ένωσης στην Ουγγαρία, ε, στην, το 68 στην Πράγα και το καθεξής. Όλα αυτά είναι μεγάλες αντιφάσεις για να μην τις αποκαλέσω και γελίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να ανακατευτώ στην συζήτηση αυτή όσον αφορά τη στρατιωτική παρέμβαση. Ο καθένας έχει την απόψή του. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να πω και μετά από τις επικρίσεις που άκουσα για την έκθεση αυτή έχω επιφυλάξεις για κάποια σημεία, αλλά έχει και ένα πλεονέκτημα. Είναι ότι τονίζει τις εξελίξεις στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα στη χώρα. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί και η κατάσταση της ασφάλειας. Χρειάζεται ένα σύστημα από τον οποίο να μπορούν να υποφεληθούν οι ίδιοι Αυγανοί. Αυτό είναι αναγκαίο. πρέπει επίσης να υπάρξει μια ειρηνική λύση. Θέλω να διευκρινίσω ότι εν μέρη διαφωνώ με αυτά που είπε ο κύριο Καν. Με κάποια άλλα συμφωνώ. Σίγουρα πρέπει να τονίσουμε το διάλογο, τη συμμετοχή των διαφόρων τάσεων και οι παστούν να συμμετέχουν επίσης, ώστε να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση σαν και αυτή στο Ιράκ. Θα υποβάλω τροπολογίες. Και θέλω να μιλήσω και για την αποναρκοθέτωση, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έχει τι περισσότερε νάρκε από οπουδήποτε αλλού. Ε. Ευχαριστώ, κύριο Σκέλαμ. Συμφωνώ ότι η έκθεση αυτή ε, είναι μεροληπτική ιδεολογικά και δυστυχώς δεν ανακλά τη θέση της πλειοψηφίας της Επιτροπής μας. Εάν θεωρεί κανείς το μεγαλύτερο πρόβλημα την παρουσία ξένων δυτικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν, τότε πώς μπορεί να εκτιμηθεί η πολιτική κατάσταση ε, σήμερα στο Αφγανιστάν. Έχουν γίνει δημοκρατικές εκλογές. Πώς θα γινόταν αν δεν είχε επέμβει η Διεθνή Δυτική Συμμαχία για να ε, κατατροπώσει τους Ταλιμπάν. Είναι εκτός πραγματικότητας η έκθεση αυτή δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Τα είπε και η κυρία Αλιομαερή πολύ ξεκάθαρα. Και καλεί σε μονομερή αφοπλισμό απέναντι σε τρομοκράτες η έκθεση. Και απολύτως ε, ξεχνάει τα ε, θύματα των Ταλιμπάν και τα θύματα της Δυτικής Συμμαχίας που ε, έπεσαν από τα πυρά των Ταλιμπάν και των τρομοκρατών. Η έκθεση βεβαίως θα πρέπει να συγγραφεί εκ νέου. Δεν χωράει βελτίωση η σημερινή της μορφή. Chairman, on a recent Πρόεδρε, πρόσφατα πήγα στο Κατάρ να δω έναν ανιψιό μου που είναι μηχανικός εκεί. Μίλησα με κάποιον Αυγανό που είναι οδηγό του. Και τον ρώτησα, τι κάνεις στο Κατάρ. Και μου είπε, δουλεύω εδώ για να εξοικονομήσω χρήματα, μετά να επιστρέψω και να σκοτώσω δυτικούς. Εγώ όμως εδώ έχω να πω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν άρχισε το 1978 με την εισβολή των Σοβιετικών. Αποσταθροπήθηκε το Αφγανιστάν. Όταν ιτήθηκαν οι Σοβιετικοί, εμείς εγκαταλείψαμε το Αφγανιστάν. Τους χρησιμοποίησαμε για να διώξουν τους Σοβιετικούς και μετά τους εγκαταλείψαμε. Γι' αυτό είναι και στην κατάσταση που βρίσκονται σήμερα. Εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να βρεθούν πάλι στη δημοκρατία και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να τους διδάξουμε, να τους βοηθήσουμε με εκπαίδευση να μπουν στο σωστό δρόμο. Είμαστε εν μέρει υπεύθυνοι για την κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Αλλά μην ε, κοιτάμε πίσω, να κοιτάμε μπροστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την έκθεση της κυρίας Λέζιν. Δεν μπορώ να συμφωνήσω ανάμεσα στο 2009 και τρία χρόνια μετά πέρασα πολύ χρόνο και έζησα στο Αφγανιστάν ως δημοσιογράφος και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είτε πρόκειται για τους Αμερικανούς είτε το οτιδήποτε η παρέμβαση αυτή δεν σταματάει τα 21 χρόνια πολέμου που ξεκίνησαν με τη Σοβιετική κατοχή και τέλειωσαν με την επίθεση του Μασούτ στους Ταλιμπάν. Το 2002, 1,5 εκατομμύριο Αφγανοί στην εξορία το κατάλαβαν και επέστρεψαν στη χώρα. Κανείς δεν τους ανάγκασε. Εκείνοι κατάλαβαν ότι 25 χρόνια πολέμου τελείωσαν και τελείωσαν χάρη σε ένοπλη παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να πω και να συμφωνήσω με τους προλαλήσατες οι οποίοι θέλουν να ξαναγραφτεί η έκθεση αυτή και να αναβληθεί βέβαια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία και έχετε το λόγο τώρα. Μπορείτε να με συμβουλέψετε για το τι μέλη γενέστε. Δεδομένων των προτάσεων που ακούστηκαν εδώ από διάφορες πολιτικές ομάδες. Ναι, μπορώ να σας δώσω την εξή συμβουλή. Να συνεχιστεί η έκθεση. Προφανώς δεν θα την αποσύρω την έκθεσή μου η έκθεση αυτή θα πρέπει όπως όλες οι υπόλοιπες εκθέσεις να ψηφιστεί εδώ στην παρούσα επιτροπή. Δεν πιστεύω ότι με μονομένες ε, ομάδες ορίζουν τι εστί πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Αυτό το ορίζουν κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι ίδιες οι ψηφοφορίες. Οπότε αυτό το δρόμο νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσουμε ε, κανονικά. Έχω όμως το δικαίωμα να απαντήσω σε μερικά πράγματα πιστεύω δεν θα φτάσω στο ίδιο επίπεδο με ορισμένα που άκουσα. Όταν μιλάει το ECR για κομμουνισμό και χειροκροτεί το σύμπαν, ε, τι συζήτηση να κάνει σε μια επιτροπή εξωτερικών. Δεν είναι πράγματα που αρμόζουν καν σε μια τέτοια επιτροπή. Μας προσάπτεται ιδεολογικά αντιαμερικανισμό. Πού το βρήκε αυτό ο κύριος Τάνοκ δεν γνωριζόμαστε και τόσο καλά για να μπορεί να το κρίνει όλες και να με αξιολογεί. Και σε εποχές κομμουνισμού ε, δεν ε, είχα και καμιά τεράστια ηλικία, ούτε ε, φορούμε από τέτοιες ιδέες. Ιδεολόγημα είναι να μην ανέχεσαι την άποψη του άλλου. Και θέλω να επανέλθω στο εξής ένας εκπρόσωπος, όχι εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος κιόλας, ε, που είπε ότι έχει μια σχέση αυρότητας με το ΝΑΤΟ, δεν βγαίνει κανένας να του προσάψει διάφορα και να βγάλει συμπεράσματα. Και ε, εγώ δεν πρόκειται να απαντήσω στο επίπεδο των δηλώσεων που άκουσα, αλλά όταν ακούω τέτοια πράγματα παρακαλώ σύντομα να μου επιτρέψετε να απαντήσω κιόλα. Τώρα δεν προλαβαίνω να συζητήσω επί της ουσίας όλα τα επιχειρήματα. Έχω την αίσθηση ότι δεν το θέλουν κιόλα οι περισσότεροι. Για μια παράγραφο που οι φιλελεύθεροι θεώρησαν απολύτως απαράδεκτη, να αναφερθώ σε αυτή, και θέλετε να τη διαγράψετε. Να σας τη διαβάσω. Ανησυχεί για τη μεγάλη εξάρτηση της χώρας από τη διεθνή βοήθεια καθώς επίσης από το μεγάλο έλλειμμα του προπολογισμού και τη μείωση των εσόδων. Θεωρεί απαραίτητο να υπάρξουν αναπτυξιακά προγράμματα έτσι ώστε η οικονομία του Αφγανιστάν όλο και περισσότερο να γίνεται ανεξάρτητη και να μην εξαρτάται πλέον ε, από ξένους δωρητές τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν και μπορούν να διαδραματίσουν σε μια τέτοια εξέλιξη τα γειτονικά κράτη. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι απαράδεκτο αυτό. Μπορώ να καταλάβω αυτά που λέτε για τις στρατιωτικές επεμβάσεις, αλλά συγκεκριμένη παράγραφος γιατί είναι τόσο ιδεολογικά φορτισμένη και πρέπει να διαγραφεί. Αυτό πραγματικά μου διαφεύγει. Ο κύριος Τάνοκ ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των γυναικών Και τον τιμά αυτό. Δεν είπα ποτέ εγώ ότι θέλω να επιστρέψουμε στους καιρούς των Ταλιμπάν. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι και σήμερα εκατοντάδες γυναίκες ε, φυλακίζονται στο Αφγανιστάν. Και σήμερα. Δείτε και ε, τα ντοκιμαντέρ του γερμανικού καναλιού ARD. Γυναίκες που θέλουν να χωρίσουν ή που θέλουν να μπορούν να περπατάνε μόνοι τους στον δρόμο. Τις συλλαμβάνουν και τις φυλακίζουν είναι γεγονός σήμερα αυτό και πρόκληση και προσπάθησα να το εντάξω στην έκθεσή μου. Έχω κάνει και προτάσεις για το πώς μπορεί κανείς να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Για τον κύριο Ντανζάν. Και το βλέπω αντιφατικό και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση να λέμε ότι είναι υπερβολικά τα χρήματα που δίνονται για ασφάλεια. Τελειώνω, τελειώνω ταυτόχρονα να ζητάμε να πληρώνονται οι άνθρωποι αξιοπρεπώς. Το ξέρω ότι είναι αντιφατικό, αλλά ισχύει. Αστυνομικοί και ε, στρατιώτες ζητιανεύουν κυριολεκτικά ε, περιφερόμενοι διότι δεν τους πληρώνουν. Και θα πρέπει ο κόσμος αυτός να ενταχθεί σε μια πολιτική ζωή. Αυτά είναι μερικά από τα σημεία που με ενδιέφεραν και έχω βάλει στην έκθεσή μου. και σε ό,τι αφορά την κατάσταση στο Αφγανιστάν, δεν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερη η δική μου θέση ή εξαιρετική. Τη συμμερίζονται πολλοί άλλοι παράγοντες και φορείς και σήμερα ε, πραγματικά είναι απαράδεκτα τα θέματα αυτά και κατωτά του επίπεδου να μου προσάπτεται ιδεολογική ε, σκοπιμότητα. Ένας κάτοικος ενό χωριού στο Αφγανιστάν έδωσε συνέντευξη για το κανάλι ARD της Γερμανίας και λέει για του ανθρώπους εδώ δεν έχει διαφορά η τρομοκρατία των Ταλιμπάν με την τρομοκρατία εκείνων που ήθελαν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία των Ταλιμπάν. Δεν το είπα αυτό. Δεν συμφωνώ απολύτω με αυτή την άποψη. Θα πρέπει κανεί να είναι αντικειμενικό ή να προσπαθεί τουλάχιστον ακόμα και αν δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όσο θα επιθυμούσε η Επιτροπή μας. Και επίσης δεν πιστεύω ότι αυτά που αυτό τον καιρό είναι συμφέρον της κυβέρνησης στο Αφγανιστάν είναι το ζήτημα που θα καθορίζει πώς θα περιγράφουμε την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα περιγράφεται μόνο με πραγματικά στοιχεία και όχι το συμφέρον της κυβέρνησης λάθη μπορεί να έχω κάνει. Υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις και διαφορετικές αναλύσεις. Τι να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Είχατε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε τη θέση σας τώρα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι ο εισηγητής οφείλει να προσπαθήσει να εκπροσωπήσει την άποψη της πλειοψηφίας της Επιτροπής και όχι την κομματική του τοποθέτηση θα πρέπει να καταβάλλεται με ΑΙ αυτή η προσπάθεια. Έχω την αίσθηση ότι εδώ υπάρχει μεγάλη πλειονότητα ε, ε, των ε, πολιτικών ομάδων που βλέπουν διαφορετικά την κατάσταση σε σχέση με εσά. Και με βάση αυτό είναι δύσκολο να υπάρξει μια συνεννόηση για μια τελική έκθεση. Και θα σας πρότεινα να ξανασυζητήσουμε στο διευρυμένο Προεδρείο τι μέλη γενέστε με την παρούσα έκθεση και τη συγκεκριμένη περίπτωση, αν συμφωνείτε. Ο κύριο Τάνοκ. Ε, Καταρχάς, αν διαβάσετε τις πρώτες τρεις παραγράφους, ε, είναι σαφές. Κοιτάξτε, δεν κάνουμε άλλη συζήτηση, αλλά... Εντάξει κύριε Πρόεδρε, αλλά από τη στιγμή που κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατο τα, οι πολιτικές ομάδες της πλειοψηφίας να συμφωνήσουν με αυτή την έκθεση δεν θα πρέπει να αναθέσουμε τη συγγραφή ε, της έκθεσης σε εσά κύριε Πρόεδρε και να ψηφίσουμε γι' αυτό και να επιτρέψουμε στην ΚΟΕ να κάνει τη δική της έκθεση ε, μειοψηφία. Ευχαριστώ. Κοίταξτε, να το συζητήσουμε αυτό στο διευρεμένο Προεδρείο και να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση και δίκαια. Ε, κύριος Μπιουτικόφερ, κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ το κόμμα μου mainstream κόμμα, πολιτική ομάδα και δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Τάνοκ. Και δεν έχει το δικαίωμα να ε, προσδιορίζει τι φρονούν ε, κάποιες άλλες ομάδες. Δεν κατάλαβα. Όλοι θεωρούν ότι τα κόμματα τους είναι mainstream, κόμματα της πλειοψηφίας. Και ε, για το ΑΕΛΚ το λέω, να έγινε και αυτό το σχόλιο. Ωραία, ξεχάστε το. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, στο διευρυμένο Προεδρείο για να δούμε. Θα είναι παρούσα βεβαίω η κυρία Λόζινγκ στι συνεδρία του διευρυμένου Προεδρείου για να υπάρξει σωστή και δίκαιη μεταχείριση. Θα ψηφίσουμε και το διευρυμένο Προεδρείο είναι ε, το όργανο το οποίο διανέμει τις εκθέσεις και που πρέπει να συζητάει αυτά τα θέματα. Και θα σας αναφέρουμε την έκβαση μετά στη συνέχεια τι θα προτείνει το διευρυμένο Προεδρείο. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στις ψηφοφορίες. The protocol to the partnership and cooperation agreement is... Πρώτα απ' όλα, πρωτόκολλο στη Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία για τη σύννεψη Εταιρική Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Ρωσία, ώστε να ληφθεί υπόψη προ χώρε τη Δημοκρατία τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να ψηφίσουμε, ναι. Εισηγητής. Ο κύριος Πρέντα. Υπέρ. Α, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Κύριος Βόλτ και τι έχει την American Express στο χέρι του. Πέρα τη οφορία. 52 υπέρ, 9 κατά, 3 αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, συστάσεις προς σχετικά με το TTIP. Ο κύριος Μιλανμόν... Όχι, ωραία, ψηφίζουμε κατευθείαν λοιπόν. Συμβασμό 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43, τροπολογία 43. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία. Το δέχεστε. Καλώς. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Θέλω να εξηγήσω ότι στα ισπανικά υπάρχει κάποιο λάθος γιατί αναφέρεται 53. Είναι 43 και για τα ισπανικά. Ναι, αλλά πάντα πάνε πιο γρήγορα οι λέει ο κύριος Μπροκ. 43 λοιπόν. Απορρίπτεται. 27 υπέρ, 36 κατά και μία αποχή. Συνεχίζουμε. 46 κατά υπέρ, υπέρ, 46 κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. 26 υπέρ, 32, 36 κατά, 2 αποχές, απορρίπτεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά άποχες έλεγχος για τις 45. Πέρας. 34 υπέρ, 28 κατά εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 59. 59. 59. 59. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 60-61. Όχι, αυτά τα καλύπτει η συμβαστική. Πάμε παρακάτω. 74 υπέρ. Υπέρ της 74. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε.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 σχεδόν τελείωσε η ψηφοφορία τώρα. Έκλεισε. Εγκρίνεται η 35 υπέρ 20 κατά και 5 αποχές.